σημείο δηλώσεις ε, της Αντιπροέδρου για τις φρικαλαιότητες στην Βόρεια Νιγηρία. κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η βία της Μποκοχαράμ στη Βορειοανατολική Νιγηρία έχει γίνει πλέον καθημερινή, πιο ακραία και πιο απειλητική για την περιοχή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συμπεριλάβατε αυτό το θέμα στη σημερινή συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό όταν συζητάμε τη δική μας ασφάλεια και τις σχετικές απειλές να μην ξεχνάμε τα όσα συμβαίνουν και αποτελούν τρομοκρατικές απειλές σημαντικές σε άλλα μέρη του κόσμου. Αποτελούν κομμάτι της στρατηγικής μας ε, επικοινωνίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τους τελευταίους μήνες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ε, άμαχοι έχουν ε, από σειρά ε, επιθέσεων και βομβαρδισμών. Η απειλή επιδενώνεται όλο περισσότερο στόχος είναι η εξάπλωση του τρόμου και η απόκτηση εδαφικού ελέγχου με αδιάκριτη στόχευση όλων χριστιανών, μουσουλμάνων, ε, θρησκευτικών ηγετών, ε, χωρικών γυναικών, παιδιών, αλλά ειδικότερα να υπογραμμίσω την επιθέση κατά χριστιανών και κοριτσιών, κοριτσιών μαθητριών ουσιαστικά, που αποτελούν σύμβολο αλλαγή της κοινωνίας τους. Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί. Σχεδόν 13.000 παιδιά από το 2009 παραπάνω από το μισό από αυτό το 2014 πάνω ε, εκατομμύρια μετατοπισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες ε, μετανάστες στο Καμερούν και στο Τσάντ που δημιουργούν εντάσεις στις τοπικές κοινότητες και δημιουργούν περαιτέρω διενέξεις. Η κατάργηση του της ένομης τάξης ε, στις περιοχές αυτές ε, καθιστά τα πράγματα πιο δύσκολα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί αλλά θα πρέπει να δεσμευτεί όλο και περισσότερο. Είναι πιο αποφασιστική για να υποστηρίξει τι χώρε αυτέ στην αγώνα κατά τη Χαράμ. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να υπογραμμίσω πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τις πληγήσεις χώρες. Βραχυπρόθεσμα χρειαζόμαστε αποτελεσματική στρατιωτική και ανθρωπιστική αντίδραση στην κρίση. Οι χώρε τη περιοχή έχουν αναλάβει να δημιουργήσουν μια πολυεθνική κοινή task force η οποία δεν έχει ακόμη κινητοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στο συντονισμό αυτής της ομάδας. Παρέχει ήδη 10 εκατομμύρια ευρώ για αντιτρομοκρατική αρρωγή στο σχετικό συμβούλιο της Νιγηρίας. Επίσης παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια για τους μετανάστες και τους μετατοπισμένους. Μεσοπρόθεσμα Επίσης παρέχουμε βοήθεια για την αναπτύξη και για θέσεις εργασίας ε, και για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Για να κερδίσουμε τον πόλεμο αυτό πρέπει να κερδίσουμε το πνεύμα και τις καρδιές των πληγέντων. Αλλιώς ε, δεν θα επιτυχούμε τους στόχους ασφαλείας και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες ε, δέσμευση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό το μήνυμα δώσαμε στον τελευταίο Υπουργικό Διάλογο με την Ιγυρία τον Νοέμβριο, που καλέσαμε την Ιγυρία να επιταχύνει την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων και να υλοποιήσει την ε, τήρηση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να μπορέσουμε να ενώσουμε μαζί τους τις δυνάμεις μας για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πιο αποτελεσματικές και πιο συγκεκριμένες. Ευχαριστούμε πολύ. Παίρναμε τώρα στους ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ομιλητής για ένα μισή λεπτό εκπροσωπεί το ΕΛΚ ο κύριος Στίερ. Ευχαριστούμε κύριε Υπετή εκπρόσωπε. Ενώ η προσοχή της Ευρώπης ήταν στραμμένη στη βάρβαρη επίθεση στο Παρίσι, στην Ιγυρία η Μπόκο Χαράμ ισοπαίδωσε την πόλη της Μπάγκα. Να επαναλάβω τα λόγια του Καθολικού Αρχιεπισκόπου εκεί Ανταδράσαμε λοιπόν τόσο ενεργά σε μια επίθεση στη Γαλλία. Το ίδιο πρέπει να αντιδράμε και όταν βλέπουμε μια τέτοια επίθεση στο Καμερούν, στην Ιγυρία ή σε άλλες χώρες. Φυσικά αντίδραμε πιο ισχυρά όταν κάτι συμβαίνει στη, δικό στη δική μας Ήπειρο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την αλληλεγγύη ολόκληρης της Ευρώπης ε, με τα θέματα του Παρισιού αλλά οι αξίες είναι παγκόσμιες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη στα θύματα του Ισλαμικού, της Ισλαμικής τρομοκρατίας στην Ιγυρία. 2.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Μπάγκα. Πρέπει να λέμε «Ζεσουή Μπάγκα» ή «Με Μπάγκα». Η Μποκοχαράμ ε, εγκαθιδρύει ένα χαλιφάτο στη Βορεια Νιγηρία και αρχίζει να αποτελεί παγκόσμια απειλή όπως οι τζιχαντιστές στη Συρία ή στη Λιβύη. Για να ολοκληρώσω, Η ερευνητική μας στόχη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή την απειλή της τρομοκρατίας. Η Μπόκο Χαράν κερδίζει έδαφος λόγω της αναποτελεσματικότητας των Νιγηριανών θεσμών. Πρέπει να βοηθήσουμε την Νιγηρία για να αναπτυχθεί σε αυτόν τον τομέα. Εκ μέρους ε, των Σοσιαλδημοκρατών για δύο λεπτά ο κύριος Νόμπετ Μόιζερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, τα θύματα της επίθεσης στην Γαλλία και πολύ σωστά ε, τράβηξαν την προσοχή μας ε, και τη συναισθηματική μας ε, συμμετοχή. Πολλοί αναφέρουν, έχουν αυτό το σλόγαν «Je suis και εγώ ξέχασα να φέρω μαζί μου ένα σλόγαν που να λέει «Είμαστε όλοι Νιγηριανοί» γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων κάτι που το αξίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Είμαστε αδύναμοι απέναντι σε όλες τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις άραγε από τη Μαυριτανία, το Μαλή, το Νίγηρα, το Τσάτι, την Νιγηρία, την Κένια, τη Σομαλία. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε στις ε, πολιτικές ελίτ αυτών των κρατών, κυρίως ε, στην Ιγυρία. Τα κράτη-μέλη βοήθησαν να εκπαιδευτούν δυνάμεις ασφαλείας στην Ιγυρία, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τουναντίον, οι δυνάμεις ασφαλείας εν μέρη λειτουργούν χωρίς ε, δημοκρατική νομιμοποίηση, χωρίς έλεγχο ε, και χωρίς την πίεση της λογοδοσίας που όλα αυτά όμως ε, εντάσσονται στην αλήθεια αν πραγματικά έχουμε κατά νου τη δράση της Μποκοχαράμ και των άλλων τρομοκρατικών ομάδων. Πρέπει να δούμε πώς θα ελέγξουμε την κατάσταση στην Ιγυρία. Τα τελευταία δέκα χρόνια 80 εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν και αυτά είναι χρήματα που τα χρειάζεται επιγόντως η χώρα για να μπορέσει να επιφέρει ε, δίκαιες συνθήκες διαβίωσης. Έχουμε μία ελίτ που ε, πλουτίζει πίζει συνεχώς ενώ παράλληλα υπάρχει ακραία φτώχεια. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι οι ε, οργανώσεις που υπάρχουν ε, στην κοινωνία, οι περιφερειακές, ε, να ενταχθούν περισσότερο στη ΜΚΟ και εμείς να τις στηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρου ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο κύριος Μπέλντερ Μπάς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχές αυτής της εβδομάδας ε, ο Αρχιεπίσκοπος Ιγνάσιος ε, Καϊχάμα αναπονέθηκε για την άγνοια της δύση για τον Μπόκο Χαράμ. Λέει, μας είπε πού είναι η αλληλεγγύη της δύση με την Ιγυρία που υποφέρει λόγω του Ισλαμιστικού ε, τρομοκρατικού κύματος. Τη Δευτέρα ο Νιγηριανός ε, Υπουργός Άμυνας είπε πως ε, έχει χαθεί ο πόλεμος εκτός εάν μας βοηθήσει μια διεθνή συμμαχία. Και οι, οι γειτονικέ χώρες, ο Νίγηρας, το Τσάντ και το Καμερούν δεν ε, είναι διατεθειμένες να παρέμβουν στρατιωτικά μέσα. Μιλάμε λοιπόν εδώ πέρα για αποσταθεροποίηση ολόκληρης περιοχής γύρω από την Νιγερία. Και χρειάζεται μια γρήγορη και στιβαρή ευρωπαϊκή απάντηση. Και να δούμε βέβαια και τις σχέσεις ε, Νιγηριανού στρατού και Μπόκο Χαράμ. Σας ευχαριστώ. Μαρίτιε Χάκε για τους φιλελεύθερους για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, η φρικτή βία των τζιχαντιστών χτύπησε και κοντά μας την προηγούμενη εβδομάδα. Και όταν ο κόσμος που πάει και ψωνίζει και δολοφονήθηκε επειδή ήταν Εβραίοι. Οι ανοιχτές ε, κοινωνίες ε, απειλούνται από τον βίαιο Ισλαμισμό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ανθεκτικοί στο να είμαστε ανοιχτοί. Αλλά όχι μόνο επιλέγουν σύμβολα της ελευθερίας έκφρασης, αλλά τα κορίτσια στην Νιγηρία, την εκπαίδευση των κοριτσιών, που είναι ο πρώτος στόχος του Μπόκο Χαράμ, που ε, κατά λέξη σημαίνει «η Δύση είναι αμαρτία». Δεν είναι δυνατόν λοιπόν το να υποχωρήσουμε μπροστά σε αυτή την βία. Το 2011 όταν ήμουν παρατηρητής προεδρικές εκλογές στην Ιγυρία σκοτώθηκαν εθελοντές σε τρομοκρατικές ε, επιθέσεις. Ε, Θελοντές που είχαν πάει να βοηθήσουν στην διοργάνωση των εκλογών και ήταν νέοι Νιγηριανοί. Τώρα έφτασαν σε νέα επίπεδα βαρβαρισμού χρησιμοποιώντας ένα παιδί για επίθεση αυτοκτονίας. Καταδικάζουμε εντονότατα αυτές τις επιθέσεις και στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε την παγκόσμια φύση της ε, τζιχαντιστικής τρομοκρατίας καθώς οι δράστες προέρχονται από όλες τις γωνίες του κόσμου και βλέπουμε πως στην Ιγυρία η τρομοκρατία έχει γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε το Ισλαμικό κράτος, την Αλκάιντα, τον Μπόκο Χαράμ και τα θυγατρικά τους δίκτυα. Ευχαριστώ. Μακάρθη για 1,5 λεπτό για την Γκουε. Ήταν συγκλονιστική η εβδομάδα στην Νιγηρία με πάρα πολλά θύματα και προφανώς λυπούμεθα τους ανθρώπους αυτούς. Και βεβαίως ε, οι πράξεις αυτές ήταν στα όρια του αδιανόητου. Πάνω από 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε λίγες μέρες, δολοφονήθηκαν και οι δυνάμεις ε, της τάξης και του στρατού δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Ήδη είπαμε πως ε, έχει και τις ευθύνες του το Νιγηριανό κράτος ε, για την κλιμάκωση και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία, παραδείγματος χάρη, πιστεύει πως τουλάχιστον 950 μέλη της Μπόκο Χαράμ πέθαναν λόγω εκτελέσεων και άλλων πρακτικών το πρώτο μισό του 2013. Τούτου λεχθέντος τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις πράξεις της Μπόκο Χαράμ που χρησιμοποιεί ένα πεδίο ως βομβιστή αυτοκτονίας, κάτι απίστευτο το οποίο πραγματικά σοκάρει και τους πιο ψημένους θα έλεγα παρατηρητές. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να δούμε τις συνέπειες ε, αυτών των πράξεων ε, σαν να συνέβαιναν οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Και ακριβώς όταν υπερασπιζόμαστε την ε, ελευθερία του λόγου πρέπει να πούμε πως υπάρχει ένα ηθικό καθήκον για να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε τη σταθερότητα και την δικαιοσύνη στην περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε έτοιμος να απαντήσετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Τζαντάσκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε Κάρθη, ε, αξιότιμοι συνάδελφε, δεν θεωρείτε ότι αυτές οι φρικαλαιότητες στην Ιγυρία οφείλονται σε ελλείψεις της κυβέρνησης της Ιγυρίας Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ε, κύκλωμα μετάφρασης. Okay. Which channel didn't work? Ποιο κανάλι δεν λειτουργούσε στο αγγλικό. Channel 2. Can you say something perhaps so that we can check whether the translation works? <laughs> Okay, sound check. <laughs> Μπορείτε να πείτε κάτι για να ελέγξουμε το σύστημα. Σωστός, μη τρέβομαι να μπόγερσκε το πρόβλημα. No, there is no English translation. Πρέπει να πω κάτι στα βουλγάρικα. Could I ask you to say something again? Πρόβα, ενώ δύο, τρία, πρόβα. Μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή, παρακαλώ. Now, Thank start again. <laughs> Колега Карти, не смятате ли, че... αγαπητέ συνάδελφε, δεν θεωρείτε ότι η ανεπάρκεια της νιγηριανής κυβέρνησης είναι ο λόγος για τις φρικαλαιότητες σε αυτή τη χώρα. Δεν θεωρείτε ότι οι διεθνείς πολυεθνικές ε, που εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους της Νιγηρίας ε, ε, πρέπει να κατηγορηθούν. Δεν θεωρείτε ότι μόνο μια στρατιωτική δύναμη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τους τρομοκράτες της Μποκοχαράμ. Δεν πιστεύετε ότι επίσης πρέπει να βοηθήσουμε ακριβώς όπως δείχνουμε αλληλεγγύη και στα θύματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Ε, ναι. Ε, κάνατε ένα σχόλιο με το οποίο διαφωνώ να λέμε ότι μόνο στρατιωτική λύση θα ήταν κατάλληλη για να αντιμετωπίσουμε την πληγή της Μπόκο Χαράμ. Ε, σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια απόκριση αμυντική, αλλά ναι, πιστεύω, ναι, οι διεθνείς επιχειρήσεις σίγουρα έχουν ε, ευθύνη και την κύρια ευθύνη έχει η Νιγηρενή κυβέρνηση. Ε, και πιστεύω ότι παντού στον κόσμο πρέπει να δείξουμε ε, πόσο συγκλονισμένοι είμαστε και εδώ και αυτό το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση των κρατών μελών πρέπει να δείξουμε το ίδιο ώστε να δείξουμε ότι είναι απαράδεκτα οι φρικαλότητες που βλέπουμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες γιατί η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολίτες ε, ε, στις χώρες μας που δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό συνέβησαν μόλις πριν από μια εβδομάδα. Για τους πράσινους τώρα η κυρία Χάταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε καθώς θρυνούμε τα θύματα αυτή τη βδομάδα της ε, σκληρής τρομοκρατικής επίθεσης στο γαλλικό τρικό περιοδικό είναι να συζητάμε αυτό το ζήτημα στην Ολομέλεια. Συμμερίζομαι όσους ε, ανέφεραν πόσο ελάχιστα προβλήθηκε διεθνώς ε, η ισοπαίδωση της πόλης Μπάγκα στη Βόρεια Νιγηρία. Αν μη τι άλλο, εδώ πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει μια διεθνής ανεξάρτητη έρευνα για να βρούμε τι ακριβώς έγινε γιατί επικύλουν και τα νούμερα των νεκρών. Φοβόμαστε ωστόσο ότι έως και 2.000 άτομα μπορεί να έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την αδιάκριτη επίθεση. Να επισημανώ ότι οι ε, Νιγηριανές ε, στρατιωτικές δυνάμεις ε, διέφυγαν καθώς συνέβαινε αυτό. Πρέπει να υποστηρίξουμε φυσικά, παρότι είναι αυτόνομη χώρα η Νιγηρία, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει επίσης να συνεργαστούμε και με την ΕΚΟΒΑ στον Οργανισμό Συνεργασίας των Χωρών της Δυτικής Αφρικής που επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Νιγηρίας, με τα μέλη της ΕΚΟΒΑ και όλους τους ενδιαφερομένους ώστε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις να λάβουν τέλος. Τέλος να επισημάνω ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι συνέβη με τα κορίτσια Τσίμποκ Οπότε πέραν το να λέμε ότι είμαστε Τσάρλι πρέπει να πούμε ότι είμαστε και τα κορίτσια Τσίμποκ και τα θέλουμε πίσω. Ευχαριστούμε. Τώρα έχουμε με τους νομιμονούς ομιλητές πρώτος Σαντιάγο Φίσας Εξέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε δώσει πολύ μεγαλύτερη σημασία σε αυτή τη σφαγή στο Παρίσι από ό,τι στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, ε, μπορώ να ξαναξεκινήσω από την αρχή. Πολύ μεγαλύτερη προσοχή αποδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης ε, στις ακραίες ε, επιθέσεις στο Παρίσι από ό,τι στη Μέση Ανατολή. Επρόκειτο για μια οργάνωση όμως στην Αφρική, Μπόκο Χαράμ, που έχει απαγορεύσει την δυτική εκπαίδευση. Από τις πληροφορίες που έχουμε, ίσως τα πράγματα να έχουν αλλάξει κάπως στην Ιγυρία. Πάντως, δολοφονήθηκαν πάρα πολύ στην τελευταία τρομοκρατική επίθεση. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να διαφύγουν. Και βεβαίως υπάρχει και το γεγονός ότι έχουμε τους ακραίους Ισλαμιστές, οι οποίοι απήγαγαν πέρυσι... Ε, 200 περίπου κορίτσια και αναφέρεται ότι μερικά εξ αυτών πουλήθηκαν ως σκλάβες και άλλα αναγκάστηκαν ε, ή προσιλητίστηκαν αναγκαστικά στο Ισλάμ. Ε, κάποια που γύρισαν στις οικογένειές τους ε, ε, είπαν ότι τα βίαζαν κάθε μέρα. Αυτό ήταν βάρβαρο και δεν νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν γρήγορες λύσεις. Αυτό για το οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο της δύση ε, πρέπει να προσπαθήσει να είναι πιο επιτυχημένη στην Αιγυρία όπως το προσπαθεί και στη Μέση Ανατολή. Αυτό που πρέπει να ενθαρρύνουμε είναι καλύτερη περιφερειακή συνεργασία, μια οικουμενική απάντηση και αυτή αυτή ε, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και από την κοινοπολιτεία. Ε, έχουμε τα ελεύθερα κράτη με την ίδια γλώσσα και γι' αυτό λοιπόν εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να επιτύχουμε θετική επιρροή από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει πολλά δικά της προβλήματα με τα οποία καλείται να ασχοληθεί. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν περνάμε στους ε, μεμονωμένους ομιλητές.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 είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, σε απόλυτη αδυναμία. Η Μπόκο Χαράμ είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διεθνής υποστήριξη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να υπάρξει αναγνώριση αυτών των δύο πράξεων και αυτές ε, να συνδεθούν με τις εκλογές ε, της 17ης και 18ης Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ κυρία Μοργκερίνη ε, που με ορίσατε επικεφαλής του εκλογικού παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρακολουθήσουμε τις εκλογές και εγώ θα προσχωρήσω σύντομα στην ομάδα που έχει ήδη συσταθεί. Αυτή η ομάδα θα ξεχωρίζει αυτή τη φορά γιατί είναι δύσκολο να ε, αναπτύξουμε τις δραστηριότητε μας σε όλη την επικράτεια της χώρας για λόγους ασφάλειας. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει είναι οι εκλογές να είναι οικουμενικές. Ε, θα αναλύσουμε την εκλογική διαδικασία και αυτό όχι μόνο κατά την ημέρα των εκλογών. Ε, θα παρακολουθήσουμε όλες τις διενέξεις που μπορούν να προκύψουν εκ των προτέρων και επιτρέψτε μου να εκφράσω μία έκκληση σε όλους να είμαστε ενωμένοι για το θέμα της Νιγηρίας. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κίνγκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Την ίδια μέρα που η Γαλλία έπλεγε από τον Ισλαμικό εξτρεμισμό έζησε η Νιγηρία τον εφιάλτη των χιλιάδων θυμάτων της Μποκοχαράμ. οποίο πεθαίνει στην Αφρική είναι θύμα του ίδιου πολέμου, της ίδιας θανατηφόρων ιδεολογίας που έπληξε την Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε την ίδια αντίδραση. Δεν υπάρχουν θάνατοι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να δείχνουμε συνοχή και ε, να δείξουμε με δύναμη ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την απειλή πριν να είναι αργά. Δεν μπορούμε να καθόμαστε αδρανείς ε, δίπλα στη σφαγή χιλιάδων ανθρώπων. Χρειάζεται μια διεθνής ε, task force με εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών οργανισμών ώστε να δώσουμε μακροπρόθεσμες απαντήσεις, δομικές. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας σημαίνει εκρίζωση των βαθιών αιτιών που οδήγησαν στη γέννησή του. Σημαίνει να καταπολεμήσουμε τον αναλφαβητισμό, τις ανισότητες, την απουσία ανάπτυξης, τα χρέη που δημιουργούνται λόγω υπερβολικής εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και να δώσουμε κίνητρα για πολιτική συμμετοχή. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγες εβδομάδες έχουμε τις προεδρικές εκλογές στην Ιγυρία. Σημαίνει να δώσουμε ένα μέλλον στα παιδιά που χρησιμοποιούνται ως όπλα Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσετε στις χώρες σας, οι χώρες σας να γίνει το επίκεντρο του κόσμου, όπως ακριβώς συνέβη στο Παρίσι. Κάποιοι από τους ηγέτες, όπως ε, επισήμανε και η κυρία Μογκερίνη, ήταν παρόντες στις 11 Ιουνίου στο Παρίσι. Ανοίξτε λοιπόν τις πόρτες σε μια ειρηνική διαμαρτυρία απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή ε, βίας κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πρέπει να λέμε είμαι η Αφρική, είμαι μπάγκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφε. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Μπονάνο. Το δέχεστε. Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Κέγκε. Αυτή η συζήτηση ήταν πολύ σημαντική για την Ιγυρία, αλλά θα ήθελα να δω μια φωτογραφία. Αυτός ο κύριος, ο ημάμιστη του Λονδίνου, ε, που λέει ότι θα πρέπει να πεθάνει ο Μωάμες ή θα έπρεπε... Ποιο κρατάει φωτογραφία του Μωάμεθ θα πρέπει να πεθάνει. Μήπως μπορούμε να μου δείξετε και εκεί τη φωτογραφία αυτού του ημάμι. Η κυρία Κέγκη έχει το λόγο. 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την άρρωστη ισλαμική ε, νοτροπία και πολιτική με τα δικά μας τα δημοκρατικά ιδεώδη. Θεωρώ ότι όσον αφορά αυτό το ερώτημα θα πρέπει να μπαίνουμε στο ίδιο επίπεδο. Εμείς δεν φοβόμαστε κανένα και πρόκειται να αποφασίσουμε με βάση την ελευθερία της έκφρασης των δικών μας αξιών να δούμε τι είναι σημαντικό και καλό για την κοινωνία μας και να αντιμετωπίσουμε αυτό το κακό, αυτό το δεινό, όπως ε, τον καρκίνο σε ένα άρρωστο. Ευχαριστώ το λόγο, κύριος Νάρτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, το πρόβλημα είναι πρακτικό, όχι θεωρητικό. Μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στην Ιγυρία, αλλά θα χρειαστούν χρόνια. Αυτή τη στιγμή μεταξύ Μπάγα και στα σύνορα Λιβύης Νιγηρίας χρειάζεται μια μισή μέρα να περάσει κανείς ο διάδρομος παροχής όπλων για τους τρομοκράτες είναι μόνο μια μισή μέρα. Οι Νιγηρανές ε, στρατιωτικές δυνάμεις είναι διεφθαρμένες. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν δυνάμεις. Η μόνη έγκυρη χώρα αξιοπιστή είναι το Τσάτ και ο μόνος τρόπος καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι η δημοκρατική βία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο τις ευρωπαϊκές δυνάμεις οι οποίες θα πρέπει να εκπαιδεύσουν, να βοηθήσουν και να σφραγίσουν τα σύνορα. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από απλά να λέμε ωραία λόγια και δηλώσεις. Θα ακολουθήσουμε κάποια συγκεκριμένη στρατιωτική πολιτική επιτόπου σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ε, χώρες. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής. Και στέλνει αλλού ειρηνευτικά στρατεύματα. Και ξέρουμε πως έχει ανισότητα, διαφθορά, γνωρίζουμε πως τα λεφτά δεν πάνε εκεί που πρέπει, ξέρουμε πως υπάρχει φτώχεια, ανισότητα και βεβαίως ε, έτσι ακριβώς ε, οι επιθέσεις αυτές οι μισογενικές ε, στα σχολεία είναι ακόμη πιο καταθλιπτικές. Αλλά υπάρχει και η απάντηση του Πρόεδρου που έστειλε συλληπιτήρια στο Παρίσι αλλά δεν είπε τίποτα για την Πάλγα. Ξέρουμε πως ε, το Μπόκο Χαράμα έχει σπάσει και τα συστήματα επικοινωνιών, αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση της ε, Νιγηρίας θα πρέπει πραγματικά να πάρει στα σοβαρά αυτή την υπόθεση. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν θα μπορέσει να ψηφίσει στις εκλογές της 14ης ε, Φεβρουαρίου γιατί είναι εκτοπισμένοι και πρόσφυγες. Χρειάζεται εδώ πέρα διεθνής στήριξη. Κυρία Λαμπέρτ, μείνετε ορθέα. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κάβερν. Παρακαλώ. Κύριε Κάβερν, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ που δέχτηκε την ε, κάρτα. Συμφωνείς με τις δικές μου ανησυχίες για το ότι δεν υπάρχει πια η διάταξη στο Σύνταγμα της Νιγηρίας που προέβλεπε εναλλάξ προεδρία μεταξύ Βορρά και Νότου και τώρα έχουμε μόνο τον πρόεδρο Γκούντλα να έλθουμε στο παλαιό σύστημα. Το ζήτημα για την εκπεριτροπής ε, προεδρία είναι ζήτημα των Ιγυριανών. Και ο ίδιος ο Γκούντλακ Τζόναθαν θα σας πει πως ε, εξελέγει άπαξ ε, και έχει δικαίωμα να είναι ξανά υποψήφιος. Εγώ θα ήθελα μια πιο δημοκρατική διαδικασία εκλογών. Χαίρομαι που υπάρχει μια αποστολή παρατηρητών για να μπορέσει να ψηφίσει ο κόσμος για να ισχύουν οι ψήφοι των ανθρώπων. Αλλά όποιος και αν βγει πρόεδρος, είτε ο κύριος Τζόναθαν είτε κάποιος άλλος, ελπίζω να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αντί να ότι δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαμπέρ. Το λόγο έχει η κυρία Βαλενσιάνο για ένα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα κορίτσι κάτω των 10 ετών έκανε επίθεση αυτοκτονίας ε, στην αγορά της Μπάγκα αφαίροντας τις ζωές πολλών τριγύρω. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το Παρίσι και να μην μιλάμε για την Ιγυρία, αλλά τι συμβαίνει και τι χρειάζεται η Ιγυρία για να καταπολεμήσει αυτή τη δολοφονική τρέλα της Μποκοχαράμ. Τι πραγματικές δυνατότητες έχουμε να βοηθήσουμε την Ιγυρία. όταν αυτοί σκοτώνουν γυναίκες ε, ε, κορίτσια χρησιμοποιούν τις αγορές ως τόπους εξασκή βίας. Όλα αυτά είναι συμβολικά. Δείχνουν ε, αυτή η δολοφονική νοοτροπία, για να την ονομάσουμε έτσι, τι προσπαθεί να κάνει στον αμαχοπληθισμό. Χρειαζόμαστε πολιτική επικοινωνία και επίγοντα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα στην έρευνα μιας πιθανής διεξόδου για αυτή την ε, ε, σημαντική χώρα της Αφρικής. Ευχαριστούμε κυρία Μίτση. Ναι. Ε, πρόεδρε. Μια ξεχασμένη σφαγή. Έτσι αναφέρθηκε στα μέσα η σφαγή στην της Μποκοχαράμ στην Μπάγκα, στην Ιγυρία είναι μια ύπουλη επίθεση της Μποκοχαράμ. Πώς θα ξεχάσουμε τα 100 κορίτσια που απήχθησαν από το σχολείο τους, που δεν πρόλαβαν να τρέξουν για να ξεφύγουν της μοίρας τους. Δεν είναι απειλή μόνο για την Αφρική αυτή, είναι και για την Ευρώπη, στο Πακιστάν και οι Ταλιμπάν εκεί ε, επιτίθεται σε παιδιά, σε σχολεία, ενώ η τραγωδία του Σαλί έβαλε την τρομοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης γιατί η Ευρώπη αγνόησε τους τρομοκρατικές οργανώσεις όπως την Μποκοχαράμ για τόσο πολύ καιρό. Πόσες άλλες ζωές πρέπει να χαθούν για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για τεράστια απειλή για τη διεθνή ασφαλεία και την ειρήνη. Οι προσθέτες απειλές αποτελούν κόκκινο συναγερμό για το μέλλον. Η Ευρώπη θα χρειαστεί να αντιδράσει αποτελεσματικά και αποφασιστικά για να υπερασπιστεί τις αξίες της κατά της τρομοκρατίας. Κυρία Γκομές, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Η κυβέρνηση της Νιγηρίας ε, δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να σταματήσει την κλιμάκωση της ε, βίας της Μποκοχαράμ ε, που απαγάει παιδιά και τα χρησιμοποιεί τώρα ως ανθρώπινες βόμβες. Η καταπολέμηση της Μποκοχαράμ δεν γίνεται μεμονωμένα. Είναι μια λερναία ύδρα κατά κάποιο τρόπο Πρέπει να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα υποστήριξης. Πρέπει στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ να αναλαβούμε κοινή συλλογική ευθύνη για να βοηθήσουμε την Ιγυρία που είναι χώρα εταίρος για να εκριζώσουμε την Ποκοχαράμ. Χρειάζεται η ΚΕΠΑ να ε, πάει την Μποκοχαράμ στο Συμβουλίο Ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Νιγηρίας με την υποστήριξη των γυροχωρών. Αποτελεί Μποκοχαράμ απειλή για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Αφρική και παγκοσμίω. Κυρία Γκομές, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Έθρειτζ. Ναι, παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. Uh, Ευχαριστώ. Μιλήσατε με πάθος για την αντιμετώπιση αυτών των σατανικών οργανώσεων και συμφωνώ. Κάτι που με ανισχύει είναι πως ακούσαμε πολλά. Συμφωνείτε μαζί μου όταν μιλάμε για προβολή της Ένωσης ε, στο σενάριο αυτό. Υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει κάποια αντίδραση και οπωσδήποτε νομίζω ισχυρότερη έλεγχη στα σύνορα με ευαισθησία θα ε, αποτρέψουν τις επιστροφές αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε πως ε, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους ε, στη Λιβύη έχουν ξεκινήσει από την Ιγυρία ακριβώς για να φύγουν από αυτό το φαινόμενο. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Μογκερίνη, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και αν θεωρούμε ότι μπορούμε να κρυφτούμε στο φρούριο Ευρώπη και αντί να πάμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, που πολεμάνε την ίδια τρομοκρατική ύδρα δηλαδή νέα ύδρα που μας δημιουργεί τα προβλήματα, είμαστε καταδικασμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Τζουφρίντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το 2009 η Μπόκο Χαράμ ανακοίνωσε την ίδρυση του Ισλαμικού Καλυφάτου στην Ιγυρία. Σήμερα ε, το 60% βρίσκεται στα χέρια τους ε, και ξέρουμε ότι τον επόμενο μήνα θα υπάρξουν εκλογές αλλά έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους που δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν και δεν τους έχουν δοθεί ακόμα τα εκλογικά ε, βιβλιάρια. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη και απευθύνεται στην διεθνή κοινότητα για βοήθεια που δυστυχώς όμως σιωπά. Πέρυσι δολοφονήθηκαν 10.000 άνθρωποι την σφαγή επίσης άλλων 2.000 ανθρώπων και ειδικά την ημέρα που γινόταν η διαδήλωση στο Παρίσι ένα κοριτσάκι με ε, δυναμικά, με δυναμίτη είχε γίνει καμικάζι χωρίς να το γνωρίζει. Τι περιμένουμε ακόμα. Η Μπάγκελ είναι μόνο η αρχή, τώρα η Μποκοχαράμ θα μπορούσε να ε, θελήσει να ελέγξει την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αφρικής με την καλύτερη οικονομία. Δεν θα περιστούν στο Τσάτ και στο Καμερούν. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήσει μόνη της και να εγκαταλείψει την Ιγυρία. Δεν αρκεί ε, να λέει κανείς «Ζεσουί Σαρλί». Επόμενος ομιλητής, κυρία Γκατζιαμπάλ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είμαι κατά οποιασδήποτε μορφής τρομοκρατικής επίθεσης και βεβαίως ε, Θέλω να συλληπιθώ τι οικογένειε των θυμάτων. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με την Μποκοχαράμ, με τις επιθέσεις στο Παρίσι. Πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχει, να ξεσπάει βία. Ο κόσμος πλήττεται από τρεις μάστιγες ε, ρατσισμός, ε, εθνικισμός και ακραίος φανατικός και ακραίος θρησκευτικός φανατισμός. Και τα τρία αυτά φαινόμενα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, τον παραλογισμό, την επιθετικότητα. Η Μπόκο Χαράμ είναι ε, μια τέτοια παράλογη οργάνωση η οποία δεν είναι προσιλωμένη στις οικουμενικές αξίες του δικαίου. Ε, δεν μπορούσαμε να εμποδίσουμε να συσταθεί η Μπόκο Χαράμ, όμως μπορούμε να εμποδίσουμε να προσχωρήσουν σε αυτήν νέοι οπαδοί. Έγινε λόγος για βραχυπρόθεσμες στρατηγικές, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική και αυτή είναι η παιδεία. Με την παιδεία μπορεί κανείς να, καταπολεμήσει, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ε, ε, τρομοκρατία. Δέχεστε μία μπλε κάρτα. Μάλιστα, τι δέχετε. Παρακαλώ, κάντε την ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την μπλε κάρτα. Μιλήσατε για το εμείς. Μήπως θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μια περιφερειακή λύση σε αυτή την τραγωδία που διαδραματίζεται στην Αφρική. Δεν θα ήταν καλύτερα όλο αυτό να το αφήσουμε στην κοινοπολιτεία και στην Αφρικανική Ένωση από το να δίνουμε τη δυνατότητα στους αντιπάλους μας να απευθύνονται και να ζητούν μεγαλύτερη βοήθεια από το εξωτερικό. Κύριε Κατήσαβάλ, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι βεβαίως και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει ε, να υπάρξει μια συζήτηση για τη δημοκρατία, αυτό είναι απολύτω απαραίτητο και βεβαίως οφείλουμε να βοηθήσουμε τις όμορες περιοχές για να προάγουν τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ε, δεν μπορούμε να αφήσουμε όμως ε, την Ιγυρία μόνη της εγκαταλελειμμένη σε αυτόν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάντα παρούσα όποτε είναι χρήσιμη. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ συμμετείχα ε, στην ε, διαδήλωση στο Παρίσι. Je suis Charlie. Ε, καταδικάζω οποιαδήποτε μορφή βία. Η Ευρώπη πρέπει να εμφανίζει ενωμένη απέναντι στη βία. Αλλά δεν είμαι μόνο Σαρλί, είμαι και Μπάγκα. Μπάγκα, η πόλη την οποία κατέστρεψαν πλήρω οι τρομοκράτε και άφησαν εκεί μετά την αιματοχυσία χιλιάδε θύματα. Η Μπόκο Χαράμ κατέχει το 70% μάλλον το 17% της Νιγηρίας και εμείς δεν μπορούμε να σιωπούμε. Οι βίες πράξεις της Μπόκο Χαράμ δεν θα εξαφανιστούν από μόνες τους. Ο λαός της Νιγηρίας μας χρειάζεται. Η Ευρώπη θα πρέπει να επιστρέψει το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης αν δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε την αιματοχυσία. Τις φρικαλαιότητες και τις πρόσφατες σφαγές στην μπάγκα της Βόρειας Νιγήριας. Ο θρησκευτικός φανατισμός οδηγεί καθημερινά την Ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ σε ακρότητες. Έτσι επεκτείνεται η επικράτεια των τζιχαντιστών στην Αφρική και δημιουργείται ένα νέο μουσουλμανικό χαλιφάτο αυτή τη φορά στην αφρική από την πόλη γκούζα μέχρι τα σύνορα του καμερούν. ταυτόχρονα οι συγκρούσεις στη βόρεια νιγηρία αυξάνουν τις μεταναστευτικές ροές προς τις χώρες της νότιας ευρώπης και την ελλάδα στην οποία χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες έρχονται μέσω τουρκίας. κυρία μογκερίνη η τουρκία έχει μετατραπεί στον κυριότερο δρόμο από όπου διέρχονται χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες προς την ελλάδα και την υπόλοιπη ευρώπη αντί να περιορίζει τις μεταναστευτικές ροές διαμέσου του εδάφους της τελικά τις διευκολύνει. ταυτόχρονα η τουρκία δεν εφαρμόζει τη συμφωνία επανεισδοχής των παρανόμων μεταναστών στο έδαφος της. τέλος η τουρκία δεν έδειξε αποφασιστική στάση κατά του χαλιφάτου του μουσουλμανικού στη συρία. είναι τυχαίο; δεν νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Καστάλντο, έπρεπε να γίνεται πολιτική συζήτηση στην Ιγυρία, να υπάρχουν σχέδια, να εκπληρώνονται ελπίδε δεδομένων των επερχόμενων προεδρικών εκλογών το Φεβρουάριο. Εδώ γίνεται προεκλογική εκστρατεία με βλήματα και με όπλα. Πολλοί κόσμος δεν θα ψηφίσει, όχι γιατί θα απόσχει, αλλά γιατί δεν, έχει, δεν είναι πια ζωντανό. Σκοτώνονται στη μέση του δρόμου, σαν να ήταν σκουπίδια. από τι αποθήκε τη Λιβύη πηγαίνουν τα όπλα στην Ιγυρία γιατί σίγουρα η Μποκοχαράν δεν τα φτιάχνει μόνη της στα δάση. Πριν μερικέ μέρε είδαμε εκατομμύρια ανθρώπου να διαδηλώνουν στο Παρίσι και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έπρεπε αυτοί οι διαδηλωτέ να αναφέρονται και στου θανάτου στην Ιγυρία και για ένα σωρό άλλα νεκροταφεία ξεχασμένα. Όχι μόνο αυτά του Σαλέμπτο. Τα συλληπιτήριά μου σε όλε αυτέ ε, τι ε, οικογένειε. Ζεσουί, Αχμέντ, είμαι Νιγηριανός, δεν είμαι υποκριτής. Το λόγο έχει ο κ. Βεντά για ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση στην Ιγυρία επιδεινώνεται και γίνεται όλο και πιο δραματική. Πάνω από 2.000 άτομα έχασαν μόλις τώρα τη ζωή τους σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση οι προεδρικές ε, και κοινοβουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σύντομα. Οι κάτοικοι της χώρας αυτής θα πρέπει να αναμένουν ακόμη και χειρότερες τώρα επιθέσεις. Γνωρίζουμε τι συνέβη στην πόλη Μπάγκα. Οι Ισλαμιστές την ισοπαίδωσαν την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο στην Ιγυρία. Ένας από τους κατοίκους της Μπάγκα έγραψε στο Twitter πώς να αισθάνομαι ασφαλής όταν ε, οι ηγέτες μας καταδικάζουν τις ε, επιθέσεις στο Παρίσι αλλά όχι τις επιθέσεις στη δική μου χώρα. Δεν μιλούν για τα θύματα στην Ιγυρία. Για αυτούς η ζωή μου δεν έχει καμία αξία. Πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα αυτή χρειάζεται ε, ε υπηρεσίες και βοήθεια δυνατή. Ευχαριστώ Για Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη. Για να αναφερθούμε και στους χριστιανούς μιλώντας για αυτή την τραγωδία, ο πρόεδρος κύριος Σούλτς ανέφερε επίσης ε, τα συλληπιτήριά του για τα 2.000 θύματα στην Πάγκα, αλλά όταν παραθέσαμε τις διάφορες διακρίσεις που μας απειλούν σήμερα δεν θέλησε να αναφέρει σε αυτό τον κατάλογο των θυμάτων ε, το μίσος κατά των χριστιανών. Το να σιωπεί για αυτό το μίσος κατά των, ε, κατά των χριστιανών σημαίνει από μόνη της αυτή η σιωπή περιφρόνηση του μίσους αυτού κατά των χριστιανών. Σας παρακαλώ να μην σιωπήσετε. Σας ξαναδίνω το λόγο κυρία Μογκερίνη για να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή την Κυριακή που ήμασταν στο Παρίσι. Σκεφτόμουν ακριβώς όπως και εσείς πως είναι και αντιπαραγωγικό να μην πούμε και να μην κάνουμε τίποτα για όσα ε, συμβαίνουν. Φαινομενικά μακριά από το Παρίσι, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολύ κοντά. Γιατί όπως είπατε πολύ, αρκετοί, αυτά τα πράγματα και πολλά από αυτά τα πράγματα συνδέονται τόσο στενά ε, έτσι ώστε δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις ε, για το ότι μπορούμε να λύσουμε μόνο ένα από αυτά τα προβλήματα και όχι τα άλλα. Και ξέρω πως τα προβλήματα του κόσμου δεν λύνονται με δηλώσεις και οφείλω να πω πως ε, έχω κάποιες αρνητικές αντιδράσεις αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ε, οι δηλώσεις είναι συμβολικές ε, και πρέπει καμιά φορά να τις κάνω εγώ και όχι κάποιος εκπρόσωπος και πρέπει να μιλάμε με την ίδια δύναμη Είτε μιλάμε για το Παρίσι είτε για την Ιγυρία και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε ότι πρέπει να δράσουμε σε διαφορετικά επίπεδα. Και βέβαια το θέμα είναι και η ασφάλεια του... και τα δικαιώματα των ανθρώπων ξεκινώντας από τα κορίτσια. Και βεβαίως είναι θέμα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που δεν θα επιτρέπει να συμβούν αυτά τα φαινόμενα και για τους ε, Νιγηριανούς βεβαίως να έχουν την ευκαιρία να έχουν ένα μέλλον στη χώρα τους. Πιστεύω πως ε, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε και το είπα στην αρχή. Είπα τι κάνουμε, είτε μιλάμε για την πλευρά της ασφάλειας, την ανθρωπιστική, δεκτή η πρόσκλησή σας να κάνουμε περισσότερα πράγματα πιθανότατα με τους υπουργούς εξωτερικών παρά με οτιδήποτε άλλο, ειδικά όταν μιλάμε για τις πτυχές της ε, ασφάλειας. Να υπογραμμίσω το εξής. Υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα είναι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνεργαστούμε εκεί με την Αφρικανική Ένωση, τον ΟΗΕ, με τρόπο συντονισμένο. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Φίσας για το σημαντικό ρόλο που έπαιξε καθώς ήταν επικεφαλής θα είναι επικεφαλής ε, της αποστολής παρατήρησης των εκλογών και θα δω τις ευκαιρίες να πω πόσο εκτιμώ ιδιαίτερα όχι μόνο την κοινοβουλευτική ε, δημοκρατία αλλά και μέσω της αποστολής αυτής της παρατήρησης των εκλογών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη διπλωματική μας δουλειά και βεβαίω χάρη στον επαγγελματισμό πολλών ε, από εσά που αφιερώνεται τόσο χρόνο και προσπάθεια γίνεται δυνατόν. Σας ευχαριστώ γι' αυτό και βεβαίως ελπίζω να σας ευχαριστήσω για κάτι ανάλογο στο μέλλον και αναμένω την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, αξιότιμη κυρία.